και τους σοσιαλιστές και δημοκρατικούς ε, κάποιες αλλαγές στα μέλη επιτροπών και διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών. Θα περιληφθούν οι αλλαγές αυτές στα πρακτικά της Συνόδου και αν δεν υποβληθούν παρατηρήσεις μέχρι την έγκριση των πρακτικών θα θεωρηθούν ως...